στην Ταϊλάνδη. Θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Τσαρνέτσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η Ταϊλάνδη είναι μια γνωστή σε όλους χώρα και μάλιστα Πολλοί έχουμε περάσει διακοπές εκεί. Είναι πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός ε, για πολλούς ε, Ευρωπαίους ε, υπηκόους. Γι' αυτό έχουμε και πολύ ευχάριστες αναμνήσεις. Αλλά δυστυχώς σε πολιτικό επίπεδο έχουμε πολύ χειρότερες αναμνήσεις και εμπειρίες. Έχουμε εδώ και δύο χρόνια πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Μετά σημαντικές ε, ειρηνευτικές διαδικασίες είχαμε την, ε, το στρατιωτικό πραξικόπημα και το στρατιωτικό νόμο. Τότε η Ταϊλάνδη ήταν από τους στήγρες της Νοτιοανατολικής Ασίας ό,τι αφορά την οικονομική της πρόοδο. Σήμερα όμως ε, θα πρέπει να ακούσει τη στεντόρια φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την έκκλησή μας ε, για επαναφορά της δημοκρατίας. Γιατί αξίζει τη δημοκρατία ο λαός της Ταϊλάνδης. Είμαι πεπισμένος και εγώ και η πολιτική μου ομάδα ότι θα πρέπει ρητά και κατηγορηματικά να μιλήσουμε για την κατάσταση στην χώρα αυτή και να επισημάνουμε στην Ταϊλάνδη ότι η οικονομική μας συνεργασία θα εξαρτηθεί από την ε, τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο λαός της Ταϊλάνδης είναι ένας φίλος λαός, ιδιαίτερα για τους Σκανδιναβούς και μάλιστα τους Σουηδούς. Για πολλούς Σουηδούς η Ταϊλάνδη είναι το δεύτερο σπίτι τους. Θα πρέπει λοιπόν ως φίλοι να μπορούμε να μιλούμε ειλικρινά μεταξύ μας, να τα λέμε στα ράντε και μεταξύ φίλων θα πρέπει να γίνονται δεκτές και κάποιες κριτικές. Η καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ ανησυχητική στην Ταϊλάνδη, γιατί ο λαός της Ταϊλάνδης αξίζει την ειρήνη, αξίζει την ελευθερία, αξίζει την ε, ελευθερία επιλογής ε, των ε, εκπροσώπων του, αξίζει τη δημοκρατία. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση προς τις Ταϊλανδικές αρχές να εξασφαλίσουν άμεση επαναφορά του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών και επαναφορά της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κοράο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο Ταρνέσκι. Όταν μιλάμε για την Ταϊλάνδη, φανταζόμαστε έναν πολύ όμορφο τουριστικό προορισμό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όμως κανείς δεν γνωρίζει σε τι πολιτικές συνθήκες ζουν οι άνθρωποι της χώρας. Μετά το πραξικόπημα υπήρξε κλιμάκωση της καταστολής των μορφών βίας, καταπίεση οποιοδήποτε, φυλάκιση οποιοδήποτε επικρίνει ή διαφωνεί με το στατικό καθεστώς. Αυτό είναι σημαντικό για τι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ταϊλάνδη και πρέπει να αποδείξουμε ότι ω Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε σε θέση να ασκήσουμε πίεση προ μια χώρα, ένα στατιωτικό καθεστώ που εμποδίζει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού μια τόσο σημαντική χώρα. Αυτό πρέπει να κάνουμε με τι οικονομικέ μα δυνάμει και πιέσει, πέραν τη διπλωματική οδού. Να προσπαθήσουμε να φέρουμε ξανά στην τροχιά τη δημοκρατία στην Ταϊλάνδη. Διότι πρόκειται για μια χώρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Παντσέρη κατόπιν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Ταϊλάνδη από καιρό ε, βρίσκεται σε μια μεγάλη πολιτική και θεσμική κρίση. Μια χώρα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προστατεύονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Θα πρέπει να δοθεί τέρμα σε αυτή την περίοδο. Δύο σημεία θέλουμε να τονίσουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να υπάρξει ένα νέο δημοκρατικό σύνταγμα για τη χώρα και να οριστεί ημερομηνία εκλογών. Πρέπει αυτή η ημερομηνία να γίνει σεβαστή από όλου ώστε να υπάρξει μετάβαση από την ε, Χούντα, τη στρατιωτική Χούντα, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση. Έπειτα πρέπει να ε, δοθεί ιδιαίτερη σημασία κυρίω των εργαζομένων, τα οποία διαρκώ ε, διακυβεύονται. Η ΟΗΕ έχει ε, εντοπίσει τα προβλήματα με τα δικαιώματα των εργαζομένων στον αλληλευτικό κλάδο και τα έχει ταυτίσει με μια σύγχρονη μορφή δουλείας. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να ε, αντιμετωπιστούν αυτές οι παραβιάσεις να μην ε, επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάψει νέα αλληλευτική συμφωνία εφόσον αυτά τα προβλήματα παραμένουν και δεν επιλύονται. Ευχαριστούμε. Ο κύριε Λοκουίλερ. Για ως 1,5 λεπτό. Η Ταϊλάνδη είναι σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, οικονομικός και πολιτικός. Οπότε θα πρέπει εμείς ως ε, φίλοι της Ταϊλάνδης ε, να αναφερθούμε στις ανησυχητικές εξελίξεις στον τομέα της δημοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν να επιστρέψει σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση και να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα. Μπορεί λοιπόν να βασιστεί στο δικό της το Σύνταγμα και στις διεθνείς τις υποχρεώσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το, την ελευθερία του συνέρχεστε. Πρέπει να σταματήσουν λοιπόν οι αυθαιρεσίες, το περιφερειακό γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα μόνο για το Μάιο του 2014 μέχρι τον Αύγουστο του 2015 κατέγραψε 1222 αυθαίρετες ε, συλλήψεις. Και μετά υπάρχουν οι λεγόμενες ε, συναντήσεις για αλλαγή συμπεριφοράς που γίνονται σε συνθήκες απομόνωσης. Επίσης υπήρξαν μέτρα κατά της ε, λαθραλίας ε, και της ε, παράνομης μετανάστευσης. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται σε ψαροκάικα, σε συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν πάρα να περιγραφτούν ως σκλαβιά. Εργάζονται ψηρά ετών χωρίς να τους πληρώνουν. Κυρίως μιλάμε για μετανάστες από την Μαλαισία, την Καμπότζη και το Μιανμάρ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λένερς για λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή είναι αποτέλεσμα της φιλίας μας με τον λαό της Ταϊλάνδης. Και άρα μία προτεραιότητα μπορεί να υπάρχει μόνο η Ταϊλάνδη να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν σε μια δημοκρατική κοινωνία με αιρετούς εκπροσώπους και πολιτική κυβέρνηση. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε να υπάρξει ένα σύνταγμα το οποίο θα βασίζεται στη δημοκρατία, την ισότητα, την ελευθερία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, γιατί εάν το σύνταγμα ε, πρέπει, αν το Σύνταγμα είναι να ισχύει στο μέλλον, θα πρέπει να περιλαμβάνει τους πάντες και ο κόσμος να έχει δυνατότητα να συμπετέχει. Βλέπουμε συχνά ανησυχητικές εξελίξεις και ζητάμε από τις αρχές να σταματήσουν όλα τα μέτρα που περιορίζουν το δικαίωμα της ελευθερίας λόγου και του συνέρχεστε και να επιτρέψουν την ελεύθερη έκφραση των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκονζάλες Πένιες. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να να ανεχθεί τις καταχρήσεις κατά στρατηγική ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη στρατιωτική κυβέρνηση της Ταϊλάνδης που εκτός του ότι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της, ε, των κατοίκων δημιουργεί απειλή της δημοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή. Ανησυχητικές είναι οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, κυρίως των μεταναστών εργαζομένων και οι καταχρήσεις ε, των εμπόρων ε, φρούτων. Έχουμε αναστείλει προσωρινά τις διαπραγματεύσει ε, για συμφωνία εμπορική με την Ταϊλάνδη. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να τη συνεχίσουμε και επίση να αναστείλουμε αμέσω και το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και να εφαρμόσουμε αυστηρά τι ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση είναι απαράδεκτη η συνέχιση τη εξαγωγή των όπλων προ μια χώρα που παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αναλάβει ε, όσον αμελητή μία πολιτική κυβέρνηση και να απελευθερωθούν ε, όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, όλοι οι πολίτες που έχουν ε, συλληφθεί από... Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στους βουλευτές εξ των ομάδων. Για το έλκο κύριο Πρέντα έχει το λόγο. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρέντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πολιτική κατάσταση στην Ταϊλάνδη έχει φτάσει σε Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου ένα στρατικό καθεστώ έχει θερπάξει την εξουσία με τη βία και παραμένει σε αυτή το δυνατό περισσότερο. Και από την άλλη έχουμε του ε, τους τη της κοινωνίας που ε, θέλει ένα δικαίωμα ελεύθερη έκφραση τουλάχιστον και ένα νόμιμο καθεστώ να αναλάβει την εξουσία. Έχει στενού πολιτικού και πολιτιστικού δεσμού με την Ταϊλάνδη η Ευρωπαϊκή Ένωση. ρόλο μα λοιπόν είναι να στηρίξουμε τη δημοκρατική μετάβαση τη χώρα και να πιέσουμε την ε, κυβέρνηση να οργανώσει εκλογές. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε ότι η διαδικασία ε, σύνταξης συντάγματος ε, θα πάρει 20 μήνε και οι πρώτε εκλογέ θα μπορούν να διοργανωθούν το 2017, δεν είναι μια αποδεκτή λύση. Χρειάζεται μια νόμιμη κυβέρνηση ώστε δυνατόν γρηγορότερα. Πρόσφατα η συντακτική συνέλευση οργανώθηκε από το Κοινοβούλιο και ε, ε, απελευθερώθηκαν κάποιοι δημοσιογράφοι. Όμω, ε, παρά τα θετικά αυτά δείγματα, οι διαφανεί και νόμιμε εκλογέ πρέπει να οργανωθούν άμεσα ώστε η ταϊλανδική κυβέρνηση να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ευχαριστούμε η κυρία Ντότζ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλωσορίζω το ψήφισμα αυτό για την κατάσταση στην Ταϊλάνδη, διότι από το στρατιωτικό πραξικόπημα το Μάιο του 2013 χιλιάδες άτομα, εκατοντάδες μάλλον άτομα έχουν φυλακιστεί παράνομα. Έχουν δοθεί υπερβολικές εξουσίες στις ειδικές δυνάμεις και πολλά ε, ε, site στο διαδίκτυο έχουν, ε, απαγορευτεί, ενώ καταπιέζονται όλες οι ελευθερίες των πολιτών θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την περίπτωση του Άντι Χολ, ενό ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίο αντιμετωπίζει ποινή 7 κάθριξη και πρόστιμο εκατομμυρίων ε, δολαρίων, γιατί έχει κάνει απλώ μια έρευνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκ μέρου μια μη ανθρωπιστική οργάνωση. Και επίση ξέρουμε και το ρόλο τη Ταϊλανδέζικη εταιρεία ε, που ονομάζεται ε, natural fruit ε, στην όλη περίπτωση του Αντιχόλ. Εδώ λοιπόν καλούμε τις ταϊλανδικές αρχές να ε, σεβαστούν τις ε, αρχές για τα, που ισχύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απελευθερώσουν άμεσα τον κύριο Χόλ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω την έκκληση να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες και καταγγελίε ει βάρο του αντιχόλου, όπω είπε η σα, Πρόκειται για ακτιβιστή των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μάλιστα είναι και Ευρωπαϊο υπήκο. Ε, θα πρέπει να στυλιτεύσουμε τι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα ο Άντι Χολ συμμετείχε σε μια έκθεση τη FinWatch το 2013 που έδειξε ότι οι καταχρήσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και οι πολιτικέ ε, ε, ουσιαστικά δουλείας ήταν ε, καθημερινότητα ενός χονδρέμπορου, τελαδού χονδρέμπορου Ανανά. Και μάλιστα ε, στις 19 Οκτωβρίου έχει νέα ε, δίκη ο Άντι Χολ και επισήθηκε σημαντική ποινή βάρος του. Επίσης ότι ότι εκπρόσωπος θα πρέπει να καταδικάσει την δικαστική παρενόχληση του Άντι και να διερευνηθούν οι καταγγελίες εις βάρος της Natural Fruit. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τον Αντιχόλ που ε, είναι πραγματικά σημαντικός ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι η Natural Fruit εξακολουθεί να στέλνει ε, φρούτα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει τις εξαγωγές της. Θα πρέπει να γνωρίζουμε την προέλευση αυτών των προϊόντων. Σας ευχαριστώ και για το ότι μείνατε εντός του χρόνου. Σόγκορ τώρα για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένουν μια ομαλοποίηση της κατάστασης στην Ταϊλάνδη αντί για στρατιωτικό καθεστώς. Καλό θα ήταν να έχουμε μια πολιτική εκλεγμένη κυβέρνηση. Και βέβαια μια κυβέρνηση η οποία θα βασίζεται στο κράτο δικαίου και την ισότητα. Επιπλέον είμαι πεπισμένος πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει τη χώρα στην διαδικασία αυτή γιατί η Ευρώπη είναι σημαντικός επενδυτής στην περιοχή. Έχουμε επενδύσει περισσότερα στην περιοχή από ό,τι η ΙΠΑ και η Ιαπωνία μαζί. Και είμαστε μετά την Κίνα ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής βεβαίως. Πρέπει να φροντίσουμε να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Δυστυχώς και κάποια χαρτιμέλη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τα τηρούν αυτά. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος η Ταϊλάνδη είναι σημαντικός εταίρος της Ευρώπης όχι μόνο στον τουρισμό αλλά και στο εμπόριο και στρατηγικό εταίρος. Και άρα με ανησυχία παρατηρούμε ότι υπάρχουν συχνά ελλείμματα στην δημοκρατία, ότι υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Συμφωνώ και εγώ με την ανησυχία για τον Άντι Χολ. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση και ελπίζω σύντομα οι Ταϊλανδικές αρχές να πάυσουν τις Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει μια ομαλοποίηση της κατάστασης και να βρει το θάρρος η Ταϊλάνδη να αποκαταστήσει την δημοκρατική λειτουργία και ίσως μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι με την εμπορική μας πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πόλσακ τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ταϊλάνδη ε, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ε, θετικές. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να καταδικάζουμε απερίφραστα αυτές τις εξελίξεις, γιατί διαβλέπουμε ένα φως στην άκρη του τούνελ. Για παράδειγμα, την άνοιξη, η ανάκληση του στρατιωτικού νόμου. Μετά την κατάργηση του στρατιωτικού νόμου, βέβαια, η στρατιωτική κυβέρνηση έχει κρατήσει παρόλα αυτά κάποια ε, εξαιρετικά έκτακτα δικαιώματα. Για παράδειγμα, προληπτικός εκφοβισμός ε, σε περίπτωση ε, που έχουμε παράνομες συναθρήσεις και 300 άνθρωποι βρίσκονται στις φυλακές εξαιτίας αυτού του νόμου. Είναι η κατάσταση, θα πρέπει να συνεχίσουμε να την παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης και να καταγγέλουμε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επαναφορά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ίσως έρθει με το νέο σύνταγμα. Ελπίζουμε τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Σας, Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη δικασία και έτσι Κάθε ομιλητής μπορεί να μιλήσει. Ο κύριος Ταραμπέλα. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, μετά το πραξικόπημα, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ταϊλάνδη διαρκώ επιθυνώνεται. Κανένα δεν το αμφισβητεί. Όποιο καταφέρεται κατά τη μοναρχία ή του σχέδιου καθεστώτο ε, φυλακίζεται ή διώκεται. Ε, οι μορφέ βία έχουν πολλαπλασιαστεί από τη στιγμή που ε, το σωτικό καθεστώ έχει αναλάβει την εξουσία και θα πρέπει να φροντίσουμε και οι στατικέ αρχές και οι αστυνομικέ δυνάμεις να επανέλθουν στη σωστή πορεία. Ε, οι στότοποι που, που επέτρεπαν ω τώρα την ελεύθερη έκπληξη των πολιτών έχουν απαγορευτεί. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπερασπιστούμε τα βασικά δικαιώματα στην Ταϊλάνδη. Επίσης, να συγχαρώ την Ταϊλανδή δημοσιογράφο που έλαβε διεθνές ε, βραβείο το 2015 για την ε, άσκηση των καθηκόντων της, των επαγγελματικών της καθηκόντων στην χώρα αυτή της Ασίας. Ευχαριστούμε κύριος Μαριάς. Για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, μετά το πραξικόπημα της 22 ης Μαΐου του 2014 που έγινε στην Ταϊλάνδη, έχουν ενταθεί οι συλλήψεις οι διώξεις οι φυλακίσεις όλων όσων αντιστέκονται όλων όσων στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. η κατάσταση πλέον είναι ε, απαράδεκτη έχει φτάσει στο απροχώρητο. μάλιστα στις 14 αυγούστου 2015 η στρατιωτική χούντα ψήφισε ένα νόμο που απαγορεύει τις δημόσιες συναθρήσεις και προβλέπεται και κάθερξη μέχρι δέκα έτη εάν κάποιος παραβιάσει αυτό τον νόμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν πρέπει να γίνεται ωρεοποίηση της το τι ισχύει στην ταϊλάνδη επειδή υπάρχουν ευρωπαϊκές επενδύσεις επειδή δημιουργείται ένας κύκλος εργασιών. πρέπει λοιπόν να αποκατασταθεί η δημοκρατία πρέπει να αρχίσουν να προστατεύονται τα δικαιώματα πρέπει να γίνουν εκλογές και κυρίως να υπάρξει και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. μάλιστα ακούσαμε καταγγελίες ότι η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της αλιείας μοιάζει με δουλεία. επομένως πρέπει να επανέλθει η δημοκρατία στην ταϊλάνδη. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Όμπερμαϊερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε πως η Ταϊλάνδη έχει φιλικούς κατοίκους και με ένα μεγάλο πολιτισμό και τα Και βεβαίως γνωρίζουμε πως έχει η κατάσταση δημοκρατία. Βεβαίως από τη μία μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όπως είπα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν κάνουμε το ίδιο για τη Σαουδική Αραβία, παραδείγματο χάρη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το τι κάνουν οι διάφοροι πολιτικοί φορείς στην ε, χώρα και να μην παριστάνουμε τον δασκαλάκο εδώ πέρα. Εγώ λοιπόν ε, ελπίζω να γίνουν εγκαίρως το 2017 όπως είναι προγραμματισμένε οι επόμενες εκλογές και να αποκατασταθεί η δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος ε, Φρουντζουλίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεδομένη τη επιδείνωση κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στην Ταϊλάνδη, όπως φαίνεται από τη λογοκρισία, σοβαρή λογοκρισία των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, την αυθαίρετη φυλάκιση και ε, σύλληψη 14 ακτιβιστών από το κίνημα της Νέας Δημοκρατίας απευθύνουμε εκκλήσεις προς τις θελανδικές αρχές ε, να απελευθερώσουν ε, όσους ε, ειρηνικά συμμετείχαν σε διαδηλώσεις. Επίσης, ο ακτιβιστής Άντι Χολ απειλείται με απειλή ευθέτους φυλάκισης και προστίμου πολλών εκατομμυρίων επειδή συνέβαλε σε μία έκθεση της Finwatch που στιγμάτιζε τις καταχρηστικές συνθήκες εργασίας από ένα Ταϊλανδό χονδρέπορα ανανά. Θα πρέπει λοιπόν ε, ε, να, βοηθήσουμε την κατάσταση για τη στη δίκη του Αντιχόλ, γιατί ουσιαστικά προσπάθησε απλώς να καταδείξει παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων στην Ταϊλάνδη. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε εδώ πέρα τώρα η διαδικασία και δίνω τον λόγο στον κύριο Επίτροπο. Sorry. Thank you, Chair. Συνάδελφοι, Συμφωνώ απολύτως μαζί σα. Η Ταϊλάνδη είναι σημαντικότατος εταίρος. Και στη σχέση με την υπόλοιπη γεωγραφική περιοχή αυτή. Ξέρουμε ότι το λαό της χώρας αυτής τον αγαπάμε για τον πολιτισμό, την οτροπία του, δεν υπάρχει όμως πρόοδος ε, στην επίλυση ενός ε, κύκλου πολιτικών αντιπαραθέσεων. Κάποιες φορές με αρκετές μορφές βίας και με συνθετικό καθεστώς. Η Ταϊλάνδη πρέπει να γεφυρώσει τα χάσματα στην κοινωνία και στα πολιτικά πράγματα. Οι γέφυρες αυτές δεν έχουν ε, ε, αντιμετωπιστεί, δεν έχουν χτιστεί ακόμη. Είναι όμως καθοριστική σημασία για την ε, υπέρβαση της κρίσης. Πρέπει να ε, δούμε πώς θα προστατευτεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πώς θα εξασφαλίσουμε μακροχρόνια δυνατότητα ανάπτυξη και ευημερία στη χώρα αυτή. Ελευθερία έκφρασης, όχι λογοκρισία. Ελευθερία του συνασπίζεστε και όχι του, του συγκεντρώνεστε και όχι κατά πίεση, καταστολή και βεβαίως ε, ελεύθερη ε, έκφραση των πολιτών και όχι βία προσεχογή στα δικαστήρια. Εδώ λοιπόν πρέπει να και να μην δικάζονται οι πολίτες από στατοδικία. Εδώ η ε, κατάσταση σωστά έχει αντικατοπιστεί στην έκθεση αυτή και σωστά το Κοινοβούλιο ζητά τον σεβασμό των ανθρωπίνων, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ταϊλάνδη και να επιστρέψει σύντομα στη δημοκρατική πορεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ήδη πολλά και θα συνεχίσει την πολιτική ε, κριτικής εμπλοκής και συστηματικής αξιολόγησης της πρόοδου της χώρας. Τα πρώτα μας βήματα ήταν να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του ΙΕ από τις 13 Ιουνίου πέρσι που ζητούν την ε, ε, ε, επιστροφή σε μια νόμιμη δημοκρατική διαδικασία για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Έχουν γίνει έκτοτε δημόσιες δηλώσεις και προσπάθεια και δουλειά για θετικές αλλαγές. Έχουμε εντείνει το έργο μας με διαφορετικές οδούς όπως διπλωματική παρακολούθηση της ε, διεξαγωγής δικών και ε, την προάσπιση όσων ε, υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Να αναφερθώ και σε ένα τελευταίο πρόβλημα που έχει να κάνει με την αισθητική κατάληψη του καθεστώτος κάτι που απασχολεί πολλούς ευρωβουλευτές και το τι γίνεται με την βιομηχανία τροφίμων στην Ταϊλάνδη. Ξέρουμε ότι τα εργασιακά στην Ταϊλάνδη είναι ένα πρόβλημα και θα φροντίσουμε να τα συνεχίσουμε το συζητούμε με τους Ταϊλανδούς συνομιλητές μας. Θετικό στοιχείο είναι ότι οι Ταϊλανδικές αρχές έχουν δηλώσει επισήμως ότι θα αντιμετωπίσουν το θέμα και θα κάνουν κάποια πρώτα επικοδομητικά βήματα, αλλά ακόμη πολλά πρέπει να γίνουν. Κανείς δεν θα έπρεπε να εργάζεται σε συνθήκε δουλεία ε, τον 21ο αιώνα. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και αγοραστές όλο και περισσότερο γνωρίζουν πως παράγονται τα προϊόντα που καταναλώνουν και απαιτούν διαφάνεια και κοινωνικώ υπεύθυνε αλυσίδε εφοδιασμού. Ε, χθες το Κοινοβούλιο στήριξε την ταχεία αναθεώρηση του πρωτοκόλου του, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά της δουλείας αυτών των μορφών εργασίας. Ελπίζω ότι η Ταϊλάνδη θα αποτελέσει ένα θετικό παράδειγμα σύντομα. Ολοκληρώνοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς ένας φίλος σε συνθήκες ε, καλές εδώ οι επικριτικές υποδοτήσεις στο Κοινοβούλιο δείχνουν ότι θα συνεχίσουμε με να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη φιλία μας με το, προς το λαό της Ταϊλάνδης, αλλά θέλουμε η κυβέρνηση της χώρας να επιστρέψει στο δυνατόν συντομότερα στην νόμιμη διακυβέρνηση της χώρας, όπως ε, αναφέρουν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2013. Τέλος, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του κυρίου Χολ, του ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συγχαίρω τους συναδέλφους που έθιξαν το θέμα. Ε, παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της υπόθεσης του κυρίου Χόλου και πολύ καιρό. Οργανώνεται αποστολή παρακολούθησης της δίκης του στις 19 Οκτωβρίου τρέχοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ε, ενημερώνεται και να εκφράζει τις ανησυχίες της στις αρχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Έχουμε λάβει 10 προτάσεις ψηφίσματος. Και βεβαίως. Ε, και 7